Παρακαλώ, καθίστε στι θέσεις σα. Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τη χθεσινής συνεδρίασης είναι στη θέση σας. Υπάρχουν ενστάσει. Όχι. Εγκρίνονται. Και προχωρώ